Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, από την Παρασκευή τα προσωπικά μας δεδομένα και η ιδιωτική μας ζωή προστατεύονται καλύτερα από τις καταχρήσεις και τη χειραγώγηση. Αυτό χάρη στην έναρξη ισχύω των νέων κανόνων για την προστασία των δεδομένων που προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτό το σημαντικό κανονισμό και κυρίως τον Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεκτ ο οποίο σύντομα θα φύγει για να γίνει υπουργό στη Γερμανία και να το ευχηθώ ότι καλύτερο. Ο Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων είναι η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση τη νομοθεσία για την ιδιωτική ζωή από τη γέννηση του διαδικτύου. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προκειμένου να εγγυηθούμε ότι οι πολίτε θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ηρεμία στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με αυτόν τον κανονισμό αποδείξαμε ότι μπορούμε να καθορίσουμε παγκόσμια πρότυπα για την ιδιωτική ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην προστασία των πολιτών παγκοσμίω και από εδώ και πέρα οι επιχειρήσεις και οι πλατφόρμες στις οποίες θα εμπιστευόμαστε τα στοιχεία μας θα πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους όταν χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας. Θα πρέπει να λαμβάνουν ρητή συγκατάθεσή μα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Δεν υπάρχει πλέον σιωπηλή συμφωνία, σκοτεινέ πτυχέ ή παραθυράκια που επιτρέπουν να παρακάμπτει κανεί του κανόνε. Οι κανόνε αυτοί θα επιτρέψουν να μην επαναληφθούν σκάνδαλα εκατομμυρίων ε, χρηστών ε, που χρησιμοποιήθηκαν τα, τους, τα δεδομένα του για χειραγώγηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση, οποιαδήποτε ε, χρήση δεδομένων θα πρέπει να κοινοποιείται με εντό 72 ωρών και προβλέπονται αυστηρές κυρώσει για εκείνους που δεν σέβονται τους κανόνες. Ακόμα και 4% του συνολικού ετήσιου ε, κύκλου, εργα... εργασίας. Για τους γίγαντες του διαδικτύου αυτό μπορεί να σημαίνει και δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον καθορισμό των προτύπων ε, για την ε, ιδιωτική ζωή, αλλά επίσης ζητά οι διαδικτυακές πλατφόρμες να είναι υπεύθυνε ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Χαίρομαι που οι μεγάλες ε, παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες δεσμεύτηκαν να σεβαστούν τους κανόνες μας. Αλλά φυσικά η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε πραγματική διακυβέρνηση ε, της ε, τεχνολογικής εξέλιξης μέσω του καθορισμού ενός κατάλληλου πλαισίου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ψηφιακής αγοράς με σαφείς ευθύνε για τους ε, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Και αυτό φυσικά πέραν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σημαίνει ισότιμο σύστημα φορολογικό και προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Επαναλαμβάνεται τώρα η συνεδρίαση του Ολομέλειας, η οποία διακόπη στι 3 Μαου. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στην ε, Ολομέλεια τη 3 Μαου έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσει. Ωραία. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας μου διαβίβασαν την